να σας πληροφορήσω ότι τη Δευτέρα μαζί με τους Πρόεδρους του Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 74 ε, ο Πρόεδρος θα υπογράψει έξι νέες νομοθετικές πράξεις. Οι τίτλοι των πράξεων αυτών θα συμπεριληφθούν στα πρακτικά της παρούσης συνεδριάσεως. Θα ήθελα όμως να καθίσετε να μην καθυστερήσουμε άλλο τις ψηφοφορίες που έχουμε. Να διευκρινίσω επίσης ότι δεν θα διαβάσω